που έρχονται από τρίτες χώρες στην Ευρώπη όπως ισχύουν και για τα προϊόντα που έχουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ.